με μικρή διακοπή γιατί δεν είχε έρθει ο Επίτροπος. Très bien. Donc nous allons commencer euh, par vous, monsieur, puisque monsieur euh, le... Έχει πρόβλημα ο εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Οπότε, κύριε Επίτροπε, έχετε εσεί το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κύριοι βουλευτέ, ο πρόεδρος τώρα πηγαίνει προ την Ιαπωνία, προς το G7 και μου είπε ο πρόεδρος να σα μιλήσω εξ ονόματο του, να σα πω ποιε είναι οι προτεραιότητε, λέει ο κύριο Κόντερς. Θέλουμε να υπάρξει κάποιο είδου ε, ανάγκη τη οικονομία παρά τη δύσκολη συγκυρία. Έχουμε 2% ρυθμό ανάπτυξη το 2015 και προ το πρώτο τρίμηνο πήγαμε παραπάνω σε ανάπτυξη από τις ε, ΕΠΑ η, ανεργία σίγουρα παραμένει σε πολλά κρατημέλη πολύ υψηλή, αλλά γενικά έχουμε πέσει σε ιστορικό χαμηλό πέντε ετία. Οπότε έχουμε πέντε εκατομμύρια περισσότερες θέσεις από το 2013. Ε, νομίζω ότι η εμπιστοσύνη ε, επιστρέφει, το βλέπουμε αυτό στους καταναλωτές, στον δανεισμό ε, και στις επενδύσεις. Θα πρέπει βέβαια να επαγρυπνούμε ε, γιατί δεν τα πάνε τόσο καλά οι εταίροι μας και πέρσι ε, είχαμε το 2009 τη χαμηλότερη ανάπτυξη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τα πήγαν καλά για δύο μέρες αγορές. Με αυτή την ε, συγκυρία που είναι αβέβαιη η ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από το τι, ε, πιθαν, ευκαιρίες μάλλον έχουμε για τον εαυτό μας. Επενδύσεις, διορθωτικές μεταρρυθμίσεις και υπευθυνότητα στη χάραξη πολιτικής. Θα πρέπει να διατηρήσουμε σταθερή πορεία. Το Κοινοβούλιο έχει σημαντικό ρόλο και Έχουμε αυτό το πλάνο για την Ευρώπη που το συμφωνήσατε ε, πάρα πολύ γρήγορα, σε λιγότερο από έναν χρόνο. Είχαμε 100 δις ε, που πήγανε σε νέες επενδύσεις και έτσι τώρα ε, έχουμε καλύτερες συνθήκες για, για νέα και δηλαδή νέες ΜΜΕ και τώρα Έχουμε τις επενδύσεις στην Ευρώπη ε, για κάποια πολύ ακριβά προγράμματα και έργα, αλλά τώρα έχουμε περισσότερα ε, τοπικά, μικρότερα, αλλά και μεγαλύτερη διαφοροποίηση, οπότε έτσι υποστηρίζονται οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ε, Το τοπικό όργανα συνεργάζονται καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και βλέπουμε αυτές τις επενδύσεις που δεν είχε καταφέρει μέχρι τώρα η αγορά με το ταμείο μας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ε, και ε, την Alzheimer, την ασθένεια, αλλά να βοηθήσουμε την άλλη μεριά και τους δανειστές γιατί στο G7 αυτό το θεματολόγιο είναι πολύ βασικό και προτεραιότητα επίσης και για την Ελλάδα. Πέρσι δώσαμε μάχη ούτως ώστε να μείνει στην Ευρωζώνη η Ελλάδα και σήμερα τα οικονομικά στοιχεία είναι καλύτερα. Επέστρεψε στην ανάπτυξη στο δεύτερο εξάμεινο του 2016 και έπεσε η ανεργία του 2015 και η κυβέρνηση ε, έφτασε σε προτιμήσεις του 0,7% του ΑΕΠ. Το πρόγραμμα σταθερότητα του Βασινού Καλογεριού έβαλε τα θεμέλια για κάποιο είδου ε, ανάπτυξη σταθερή και τώρα εξασφαλίστηκε η θέση της χώρας στην Ευρωζώνη. Έχουμε τώρα την πρώτη αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο σας λέω, ότι άρχισε τώρα η κάλυψη του χρέους και αυτό δικατοτρίζει τις προσπάθειες όλου του ελληνικού λαού και σήμερα είναι δυνατόν να κάνει μια θετική στροφή πορείας η Ελλάδα, οπότε θα έρθει και η ώρα των ξένων επενδυτών. Στα πλαίσια του G7, πάντοτε εμεί προσπαθήσαμε να έχουμε παγκόσμια οικονομία, να διέπεται από κάποιου κανόνε, να υπάρχει συνέχεια περισσότερη διαφάνεια και να είναι τα πράγματα όσο γίνεται πιο ε, δίκαια. Προσπαθούμε να εξαγάγουμε στην παγκόσμια αγορά τις καλύτερες πρακτικές μας και σε αυτή τη συνάντηση θα συνεχίσουμε και μαζί με τους εταίρους του G7 εμείς ε, θέλουμε να αποδείξουμε το ότι το παγκόσμιο εμπόριο μπορεί να ωφελήσει τους πάντες, όχι μόνο ε, όλες τις χώρες αλλά και όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε, βέβαια βραχυπρόθεσμα υπάρχουν οι κερδισμένοι και οι χαμένοι. Αυτό είναι το επιχείρημα των λαϊκιστών παντού, αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε πιο δίκαιους κανόνες του παιχνιδιού, να τηρούνται οι κανόνες αυτοί και άλλα επίσης να δείξουμε ότι μακροπρόθεσμα θα υπάρχει ευημερία με ανοιχτή στάση και με σύστημα εμπορικών συναλλαγών. Πέρσι ήμασταν οι πρώτοι όσον αφορά τη διαφάνεια στα φορολογικά. Τώρα έχουμε αυτή τη συμφωνία για τις φορολογικές ρυθμίσεις και έχουμε και το σύστημα της έκθεσης αναχώρα. Το μήνυμα μας είναι σαφές. Όλοι θα πρέπει να πληρώνουν αυτό που τους αναλογεί σε φόρους και θα πρέπει σε συνεργασία με το G7 να εξασφαλίσουμε ότι πρόκειται για μια πραγματικά παγκόσμια προσπάθεια. Συμφώνησαν τα κράτη-μέλη να έχουν αυτά τα κεντρικά μητρώα για τον beneficial ownership, την, τον τελικό δικαιούχο, τον πραγματικό δικαιούχο, οπότε θα πρέπει ε, να μην μπορεί κάποιος να φοροδιαφύγει και θα πρέπει να είμαστε επίσης αυτοί για όσους ε, παραβάλλουν τους κανόνες και ελεύθερο εμπόριο να σημαίνει δίκαιο εμπόριο. Σας διαβεβαιώνω σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα στεγανό σύστημα άμυνα εμπορική και αν κάποιο τρευλώνει την αγορά, εμεί αναλαμβάνουμε δράση. Έχουμε ρεκόρ όσον αφορά ε, το dumping για την χαλιβουργία και είπαμε και με το, στο G7 ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, προτάσεις ούτως ώστε να μην έχουν περπαραγωγή και να υπάρχει εποπτεία διεθνής ούτως ώστε όλοι διεθνώς να συμμορφούνται. Και για να δούμε τώρα τι γίνεται με το προσφυγικό. Κάτι το οποίο επίση έχει προτεραιότητα στο θεματολόγιο του G7. Είπε η Επιτροπή ότι ευθύ εξ αρχή μόνο οι παγκόσμιε λύσει θα αποδώσουν. Και ε, εν προκειμένου βοηθήσατε ούτω ώστε να έχουμε μια πανευρωπαϊκή στρατηγική, σφαιρική, να σώσουμε τον κόσμο που διασχίζει τη θάλασσα, ανθρωπιστική βοήθεια, ε, προστασία των συνόρων, να βοηθήσουμε τις χώρες που επιέζονται με την κατάσταση και επαναπατρισμό και από την άλλη μεριά να καλύψουμε τους ετούντες άσυλο και το 2015 αλλά και το 2016 Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έδωσε πάνω από 10 εκατομμύρια για την κρίση του προσφυγικού και μεταναστευτικού. Οπότε με αυτή τη στρατηγική θα έχουμε το περιθώριο να μπορέσουμε να ενατενίσουμε το μέλλον και μαζί με τους εταίρους μας θα πρέπει να έχουμε τη σωστή ε, ανταπόκριση και αντίδραση και να αντιμετωπίσουμε τις ε, ρίζες του προβλήματος. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε κάποια εναλλακτική ε, στους όσους ζητούν άσυλο και να μην ρισκάρουν τη ζωή τους και πρόκειται για τον καλύτερο τρόπο να καταπολεμήσουμε τους διακινητές και επίσης να ξανααποκτήσουν αξιοπρέπεια αυτοί που πραγματικά χρειάζονται την προστασία μας για το ενεργειακό. Από τη Συμφωνία του Παρισιού είναι προς τώρα αρχίζει το έργο μας, εξημισμό της οικονομίας και αλλαγή του μοντέλου κατανάλωσης και παραγωγής. Οπότε χρειάζονται νέα κίνητρα ε, για όλες μας τις πολιτικές. Το μήνυμα είναι σαφές, αλλάζει το επιχειρηματικό μοντέλο για τις βασικές μας επιχειρήσεις, νέες ε, δεξιότητες, νέες ε, ε, διαδικασίες και θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε τη φιλοδοξία να γίνουμε πρωτοπόροι όσον αφορά τα ανανεώσιμα. Έχουμε τώρα ένα εκατομμύριο ε, θέσεων εργασία και 130 δισεκατομμύρια τζίρο ετησίω. Οι ευρωπαϊκέ εταιρείε σήμερα είναι το 40% ε, του, του, του, όλου τοπίου των ανανεώσιμων. Έχουμε ακόμα προβλήματα. Το 2013 παντού είχαμε κάποιε επιδόσει για το ρητά καύσιμα που φτάνουν στα 500 δις ευρώ. Μιλάμε για πολλά χρήματα τα οποία πήγαν στο λάθος μέρος. Το G7 υπό τη Βαθμία θα καταργήσει αυτές τις επιδοτήσεις μέχρι το 2025. Οπότε θα πρέπει και το G20 να υιοθετήσει το ίδιο μέτρο. Επίσης χρειάζεται συντονισμός και θα πρέπει να δοθούν ε, λύσεις παγκόσμιες όπως για το μεταστατικό έτσι και για την οικονομία. Και εμείς αυτό θα πρεσβεύουμε. Να έχουμε παγκόσμια οικονομία που να την διέπουν κάποιοι κανόνες. Ανοιχτή κοινωνία, έτσι θα πάμε προς την ασφάλεια και προς την ευημερία και ε, σήμερα σε αυτόν τον αβεβαιό κόσμο αυτή μας η συμβολή έχει βαρύνουσα σημασία. Σας ευχαριστώ και τώρα θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ράντζελ. Ένα λεπτό εξ ονόματος του Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να καλησπέρισω τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς και θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι σαφές ότι η ατζέντα του G7 είναι τεράστια. Η Ιαπωνική Προέδρια δεν δίστασε καθόλου να βάλει στην ημερήσια διάταξη όσο πιο πολλά μπορούσε. Σε τέσσερα σημεία θα ήθελα να εστιαστώ. Καταρχά, οι επενδύσει. Εδώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλει μια προσπάθεια. Το σχέδιο Juncker δεν επαρκεί, πιστεύω. Οι μεγαλύτερε οικονομίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία έχουν καταθέσει ιδέε και θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Κάποιες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ε, μεγάλες επενδύσεις που θα επιτρέψουν να προχωρήσει η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, όπως είπε ο πρόεδρος Ομπάμα πρόσφατα, είναι, το σημαντικό είναι οι χώρες του G7 να χρησιμοποιήσουν ε, τις δυνατότητες που έχουν. Δεύτερο θέμα που επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα τα δημοσιονομικά, τα φορολογικά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά του φορολογικούς παραδείσους. Πρέπει να κάνουμε πιο πολλά πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή και εδώ είναι μεγάλη ευθύνη του G7 και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι άλλες του G7 θα συμμετέχουν σε ό,τι αφορά την προσφυγική κρίση. Η Ιαπωνία, η Αυστραλία δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Τέλος, ένα άλλο βασικό ζήτημα για μένα είναι το θέμα του ιού Ζήκα. Ακούμε πολλά για τον ε, έμπολα, αλλά ο Ζήκα ήδη έχει φτάσει στο νότιο τμήμα της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αποτέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Τσάνι. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε, αξιότιμε, είπατε ότι η οικονομία θα πρέπει να λάβει την απαραίτητη έμφαση. Δεν πιστεύετε όμως ότι η εκδήλωση αυτή του G7 αποτελεί μια μονητική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους άλλους φορείς και παράγοντες ότι χρειάζεται αλληλεγγύη αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το θέμα για παράδειγμα της προσφυγιάς αποτελεί δικό μας θέμα. Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης του θέματος της αλληλεγγύης στα πλαίσια του g Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή που μου θέτετε. Εγώ ουσιαστικά αυτό που είπα είναι το εξή. Σε ό,τι αφορά θέματα οικονομικής ανάκαμψης, οι πιο αναπτυγμένες χώρες έχουν υποχρέωση επένδυσης και βοήθειας. Παροχής βοήθειας προς τις πιο δυναμές χώρες. Αυτό ισχύει σε παγκόσμιο αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό είμαι βέβαιος ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό από μόνη της. Θα πρέπει να μας βοηθήσουν γιατί πολλά μπορούμε να κάνουμε και πολλά κάνουμε, αλλά υπάρχουν ισχυρές χώρες που θα πρέπει και αυτές να μας βοηθήσουν. Θα πρέπει και αυτές να λάβουν τις ευθύνες τους. Ευχαριστώ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, κυρία Μόσκα σε αυτή την ε, ιστορική συγκυρία η παγκόσμια συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί και να δώσει αποτελεσματικές απαντήσεις. Μία μεγαλύτερη ε, ε, παγκοσμιοποίηση καλύτερη από αυτήν που έχουμε είναι η μόνη απάντηση για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ιδέες που θεωρούσαμε ότι είχαμε ξεπεράσει εθνικισμός, ξενοφαβία ρατσισμός. Ελπίζουμε λοιπόν να είναι πάρα πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα του G7 και τα ίδια να είναι και τα αποτελέσματα από τη βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι την ενέργεια. Ένα σημαντικό στοιχείο θα είναι το διεθνές εμπόριο το οποίο ε, πρέπει να σταματήσει τους ε, ε, δασμολογικούς φραγμούς και μη δασμολογικούς φραγμούς και να προσφέρει ισότιμους όρους σε όλους. Βάσει και του ψηφίσματος που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από δύο εβδομάδες, ελπίζουμε να βρούμε ένα τρόπο συνεπού σχέση με την Κίνα, που είναι σημαντικός εταίρος, αλλά πρέπει να συμμετέχει και αυτό στον καθορισμό ενός δίκαιου και βιώσιμου εμπορίου κυρίως όσον αφορά το καθεστώς της ε, οικονομίας ε, κλίμακας ε, που θέλουμε να δώσουμε στην Κίνα και κυρίως με τα όσα γίνονται για τον Καχάλιβα και το σεβασμό των κοινών κανόνων για την πρόσβαση στην αγορά. Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε με ικανοποίηση το σημείο για την ισότητα των φύλων στην ημερήσια διάταξη του G7. Πάντα το θέμα της ενδυνάμωσης των γυναικών μας απασχολεί και ελπίζουμε με την ευκαιρία του G7 να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις ανοσότητες ε, των φύλων με συγκεκριμένα μέτρα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του ECR για 1,5 λεπτό κύριο Χένκελ. Κύριε Αντιπρόεδρε, πάνω πάνω στην ατζέντα του G7 είναι η παγκόσμια οικονομία και δικαίως για, τα, για τους εξής λόγους. Καταρχάς, η παγκόσμια οικονομία σήμερα δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα όσο παλιά και αυτό πλήττει και θα πλήξει κυρίως τις χώρες του τρίτου κόσμου. Κατά δεύτερον, ο μεγαλύτερος κινητήριος, ε, κινητήρια μηχανής της, εθνικής, της ε, παγκόσμιας οικονομίας, η παγκόσμια οργάνωση ε, αυτή, δεν πάει καλά. Και κατά τρίτον, η Ευρωζώνη δεν τα πάει καλά εδώ και καιρό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τον πρόεδρο Τούσκ και Γιούγκερ σε ό,τι αφορά και την Ιαπωνία. Καταρχάς να κάνετε μία νέα αφετηρία σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο εμπόριο. TTIP, ZETA και TPP. Η παγκοσμιοποίηση, ξέρετε, δεν είναι μόνο οικονομικό φαινόμενο. Δεν έχει να κάνει μόνο με προϊόντα και οι υπηρεσίε τις οποίες διακινούμε σε όλο τον κόσμο έχει να κάνει και με τη δημοκρατία και άλλες αξίες. Κατά δεύτερον, το γλυκό δηλητήριο μιας υποτίμησης να το κοιτάξετε και κατά τρίτον θα σας ρωτήσουν σίγουρα γιατί έχει τέτοια προβλήματα τα τελευταία χρόνια η Ευρωζώνη. Η απάντηση είναι το one size fits all. Τα νομίσματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην οικονομική πραγματικότητα. Θα πρέπει να σταματήσουμε να υπόκεινται όλα αυτά στην, στο νομίσματα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μπλε κάρτα, λέει η Πρόεδρος. Την αποδέχεστε από τον κύριο Κασπάρη. Έχετε το λόγο. με κύριε Χένκελ, αναφερθήκατε στα θέματα της Ευρωζώνης. Πιστεύετε ότι η Ευρωζώνη το πρώτο τρίμηνο είχε μεγαλύτερη ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του έτους από ό,τι της είπα. Αυτό μήπως θα μπορούσε να σας κάνει να ξανασκεφτείτε τα πράγματα σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη, αν λάβετε υπόψη για την πραγματικότητα που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Κοιτάξτε, ε, στην πραγματικότητα συγκαταλέγεται και η άλλα αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι μόνο οι 90 ημέρες αυτές που αναφέρεται. Εγώ αναφέρομαι σε 10 χρόνια και αυτά τα αναφέρει και στα στοιχεία του ΆΣΑ. Φαίνονται ξεκάθαρα. Πίσω από τα είπα, πίσω από τον υπόλοιπο κόσμο βρισκόμαστε στην Ευρωζώνη και πίσω και από τις υπόλοιπες χώρες που δεν έχουν ευρώ. Ευχαριστώ ο κύριος Τελίσκα από τους Φιλελεύθερους. Δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, Καταρχάς να σας πω ότι η Ολλανδική Προεδρία σαφέστατα δεν προσδίδει τόσο μεγάλη σημασία στην σύνοδο του G7, αλλά χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της προσδίδει και συμφωνώ με πολλά από όσα είπατε κύριε Αντιπρόεδρε. Υπάρχουν μια σειρά από σημαντικά θέματα, θέματα τα οποία έχουν σημασία για την ημερήσια διάταξη, σημασία ε, ε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να επιδείξει λόγω και όλων των κρίσεων που έχουμε αντιμετωπίσει και υπάρχουν αρκετά θετικά μηνύματα ε, και τα θίξατε κι εσείς. Με χαροποίησε αυτό που άκουσα και για τις επενδύσεις, τις διερθρωτικές μεταρρυθμίσεις και φυσικά τα υγιή οικονομικά. Ε, όσον αφορά τη στρέβλωση της αγοράς και την ε, στάση που πρέπει να τηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ε, χρησιμοποιήστε και τον όρο εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη στις αγορές. Εγώ τον όρο εμπιστοσύνη θα τον χρησιμοποιούσα σε διαφορετικό πλαίσιο, εμπιστοσύνη στο G7. Πιστεύω ότι η πραγματικότητα είναι ότι από τις τελευταίες συνόδους του G7 δεν είχαμε και τόσα πολλά για τα οποία να μπορούμε να χαρούμε. Το G7 για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό φόρουμ και σίγουρα θα μπορεί να είναι κάτι πολύ επιτυχημένο. Αλλά υπάρχουν κάποια ουσιαστικά στοιχεία. Να εντοπίζονται τα προβλήματα, αναφέραμε κάποια εξ αυτών και υπάρχουν και αρκετά προβλήματα. Ε, κατόπιν πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε κάποιο βαθμό συνένεσης, αν όχι σε ομοφωνία. Και αυτό φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτό με φέρνει και στο τρίτο συστατικό, το οποίο είναι ουσιώδε και ίσω θα μπορούσε να είναι και καλή ε, περίπτωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εν γέννη να αναλάβουμε τα ενία. Αυτό το οποίο λείπει, αυτό το οποίο ειστερεί το G7 τα τελευταία χρόνια είναι η κατάλληλη ηγεσία. Ε, είναι πραγματικότητα αυτό. Και αν δούμε το, την ημερήσια διάταξη, είναι πλήρη η ημερήσια διάταξη, είναι πολύ εύστοχα τα θέματα, αλλά γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι σίγουρα δεν θα συμφωνήσουμε στι κοινέ ε, στρατηγικέ ανάπτυξη. Δεν θα συμφωνήσουν οι υπουργοί. Μπορεί να είναι καλύτερη βέβαια η σύνοδο, αλλά ένα από τα ουσιαστικά ζητήματα τη ημερήσια διάταξη ξέρουμε εκ των προτέρων ότι δεν θα μπορέσουμε να το συμφωνήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να προτρέψω τον πρόεδρο Γιούγκερ και τον πρόεδρο Τούσκ να επιδείξουν τον ηγετικό τους ρόλο και να μην στεκόμαστε στο περιθώριο. Να είμαστε περήφαμοι, να αναλάβουμε τα ημεία και να έχουμε αποτελέσματα. Αποτελέσματα περιμένουν από μας. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Φρουντζούλικα για σας. Δέχεστε. Ο κύριος Φρουντζούλικα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, Ξέρετε ότι η αλλαγή του κλίματος είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για το μέλλον μας και έχει σημασία και με, για τους μετανάστες που έρχονται κυρίως από την υποσαχάρη Αφρική. Δεν πιστεύετε ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να αναλάβει τα ενία στην ε, σύνοδο του G7, διότι αναφερόμαστε στην εμπιστοσύνη και να ζητήσει από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 7 χωρών να κυρώσουν το συντομότερο δυνατόν τη Συμφωνία των Παρισίων για να αποτελέσουν και το παράδειγμα για τις άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ. Ναι, αξιότιμε συνάδελφε, αναφέρθηκα σε ηγετικό ρόλο και νομίζω ότι είναι συνολικός αυτός ο ρόλος. Όλα αυτά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι σημαντικά. Αλλά επίσης αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να καταλήξουμε και συμφωνία σε διάφορα ζητήματα. Η ηγεσία δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ε, θα είναι κάποιος πολύ μπροστά ενώ οι υπόλοιποι θα υστερούν. Και όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, ναι, μεν είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα, αλλά χρειαζόμαστε μια παγκόσμια συμφωνία και να προσπαθήσουν όλοι για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκονσάλε Πένιας για ένα λεπτό εξ ονόματος τη ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι προβληματιζόμαστε όσον αφορά την τοποθέτηση της ε, Ένωσης, όσον αφορά την οικονομική στρατηγική ε, κόντρα σε αυτήν την αυξανόμενη αβεβαιότητα για τα οικονομικά όλου του πλανήτη. Βέβαια θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το φόρουμ ούτως ώστε να σταματήσει η κερδοσκοπία, να καταπολεμήσουμε τους φοροπαραδείσους και ότι υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα η οποία τώρα ε, γίνεται από τις ελίτ και ε, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει τίποτα, υπάρχει κρίση όσον αφορά τις επενδύσεις και εκείνοι που έχουν πληγεί περισσότερο είναι οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες από τις μεγάλες δυνάμεις που συνεχίζουν να βοηθούν την ε, κερδοσκοπία και ε, θα έπρεπε να βρουν λύσεις για την καθημερινή ζωή και έχουμε τα πλάνα Juncker αλλά πάντοτε βοηθούν αυτούς που βοηθούσαν ναι, πάντοτε και όχι αυτούς που θα έπρεπε να βοηθούν. Άρα θα πρέπει να γίνει κάτι πέρα από την μιζέρια και από ε, την ε, λιτότητα. Και ούτε το, το TTIP δεν αφορά το, τον κοσμάκι, αλλά αφορά τις ε, πολυεθνικές αυτές ωφέλη. Γκίγκολτε, ένα μισή λεπτό για τους πρασίνους. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε Δύο σημεία θα ήθελα να δείξω. Στο G7 πριν από ένα χρόνο το μεγάλο θέμα ήταν η απανθρακοποίηση. Για την, ε, να καταστεί η παγκόσμια οικονομία πιο φιλική προς το κλίμα και παράλληλα να δώσουμε και μια οικονομική όθηση. Το είπατε και εσείς ο ίδιος. Παράλληλα είναι οι ίδιες οι χώρες αυτές που μαζεύονται και εξακολουθούν να επενδύουν σε άνθρακα, πατρέλαιο κτλ. Συνεχίζονται αυτές οι επιδοτήσεις στις βάρος του περιβάλλοντος. Τι κάνουμε στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Υπάρχει κάποια πρόταση για όλα αυτά. Για να τερματιστούν αυτές οι επιδοτήσεις που βλάπτουν το περιβάλλον. Στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, ανταυτού, βλέπω μείωση της ενίσχυσης των οικολογικών πολιτικών αντί για ενίσχυση τους. Δείξτε λοιπόν τόλμη στον τομέα αυτό και το G7 θα πρέπει να πραγματοποιήσει αυτά που είχε προεξαγγείλει. Κάτι άλλο. Πριν από δύο μήνε ψηφίσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο την έκθεση Γκουλάρ, ζητήσαμε πιο αυστηρού κανόνε σε περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων για την, ε, το καθήκον λογοδοσία σε ό,τι αφορά τις παγκόσμιες αυτέ τα παγκόσμια θεσμικά όργανα θα παρουσιάσετε αυτές τις προτάσεις στο G7 και πώς θα πραγματοποιήσει το G7 τις προτάσεις αυτές. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόσει στις εργασίες της τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω μία απάντηση. Ευχαριστώ ο κύριος Οφλίν για δύο λεπτά από το EFTD. Ευχαριστώ. Η πραγματικότητα είναι ότι η Επίτροπη δεν θα πάνε στην πιο σημαντική συνάντηση στο G7 θα είναι δηλαδή η, η προειδοποίηση που παγώνει το αίμα υποτίθεται των Βρετανών να μην ψηφίσουν υπέρ του Brexit. Ε, οπότε ε, θα είναι αντιπαραγωγική η παρουσία των επιτρόπων ε, ώστε να κάνουν το σωστό η Βρετανία για να αντιμετωπίσουν την αποτυχία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό δεν είναι γελίο ότι θα πρέπει να βρουν κάποια δικαιολογία για, το, για την αποτυχία του στα οικονομικά γιατί βλέπουμε μας, μας λέτε τώρα ότι παρά το ότι παντού όλο πάνε στραβά στην οικονομία εσείς έχετε ε, ανάκαμψη ωραία αυτά που λέτε αλλά ε, τα, τα φάξιτ λένε ότι ακόμα υπάρχουν ε, κάποιες επενδύσεις που είναι πολύ χειρότερες από πριν την από ό,τι πριν την κρίση. Η οικονομία μας είναι για την εντατική. Το 2008 ξεκίνησε η κρίση, ακόμα δεν έγινε ανάκαμψη. Και λέτε ότι θα, ε, το 2017 θα έχετε 10% για την ανεργία. Όλα αυτά είναι ψευδής πόθη, δεν είναι ε, ενημερωτικά. Οπότε, ε, όπως λέγανε στο σινεμά, θα είμαστε εκατομμυρίουχοι τέτοια εποχή, αλλά το θέμα δεν είναι η Ευρωζώνη να δώσει τη μάχη της στη, στη διεθνή σκηνή, αλλά αυτό το οποίο κάνουμε είναι να είμαστε βαρύδι για την παγκόσμια οικονομία. Και τώρα επομένω ψάχνετε συνέχεια ε, για το, το επόμενο G7 του 2017 ε, αλλά τελικά το ευρώ ήταν η θραντική ποινή για την ε, ανάπτυξη. Λεμπρετών Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η ιστορία ε, τελικά έκανε το, το, αστείο να πάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί και στο G7 που είναι κράτη και στις 26 και 27 επομένως θα γίνουν αυτά στην Ιαπωνία. Δυστυχώς θα είναι αρνητική η επίδραση όσον αφορά τη λύση των τριών προβλημάτων που θα ζητηθούν από πλευράς οικονομικής είπατε ότι πάλι θα οδηγηθείτε σε έναν ε, αχαλήνοτο φιλελευθερισμό. Πρόκειται για ε, ε, συνέχιση των περσινών συζητήσεων. Δεν ακούτε τις ανησυχίες του κόσμου. Τώρα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική πρόκειται να επιτεθείτε στην Ρωσία αλλά η Ρωσία αντικειμενικά είναι ο βασικός μας σύμμαχος κατά των Ισλαμιστών και κατά των τρομοκρατών. Τώρα όσον αφορά το μεταναστευτικό πρόκειται να μην κάνετε πάλι τίποτα καινούριο. Δεν θα βρείτε κάποια λύση, γιατί η λύση είναι να υπάρξει βοήθεια σε επίπεδο παιδείας και οικονομικής ανάπτυξης σε εκείνες τις χώρες που το χρειάζονται, ούτως ώστε να κρατήσουν τον κόσμο στην χώρα τους. Αλλά δεν σας νοιάζει. Τώρα ε, στις 24 Μαΐου ε, είπαμε ότι έχουμε την συνάντηση ε, ε στην συνάντηση την ανθρωπιστική, αλλά δεν πήγατε εκεί πέρα. Κύριε Λεμπρετό, ο κύριος Κούντερς είχε πρόβλημα, αλλά θα έρθει. Υπάρχει μία, μία κάρτα μπλε από τον κύριο Τζαμπάσκι. Αποδέχεστε, μάλιστα, Τζαμπάσκι. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Λεμπρετόν. η ηγέτες στο G7 συμφώνησαν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Θεωρείται ότι είναι απαρχαιωμένος θεσμός το G7 και ότι δεν βοηθάει σήμερα γιατί όλο ένα και ανέρχεται η Κίνα και η Ινδία. Μήπως έχουμε κάποια επικάλυψη αυτών των θεσμικών οργάνων με το G7. Κύριε ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα ερώτησή σας. Νομίζω ότι το G7 είναι ένας θεσμός ενδιαφέρον. Μπορεί να βοηθήσει όπως και άλλοι θεσμοί στην επίλυση των διεθνών προβλημάτων. Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφορίας, ε, βέβαια και χρειάζεται για πολλούς τομείς και για την καταπονόμηση της τρομοκρατίας. Εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο πρεσβεύει την συνεργασία των κυριάρχων κρατών. Συμφωνώ με την ανταλλαγή πληροφοριών. Αρκεί να μην βάζει χέρι σε αυτά τα στοιχεία η Επιτροπή των Βρυξελών που τελικά ματαιώνει οτιδήποτε καλό ε, πρόγραμμα υπάρχει ιδέα. Μπάλτσο. Θα πρέπει να νιώθουμε ικανοποιημένοι γιατί στο θεματολόγιο του G7 θα συζητηθεί το μεταναστευτικό. Και ε, μας εξήγησε ο κύριος Αντιπρόεδρος ότι πρόκειται για ένα μέτωπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους παγκοσμίω. Τι εννοείται όμως, μιλάτε για τα οικονομικά και μιλάτε για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς, αλλά τι θα κάνουν οι εταίροι μας από όλο τον κόσμο, τι θα κάνουν οι ΙΠΑ, Η Αραβική Άνοιξη προκλήθηκε από την εξαγωγή των όπλων από εμά. Να, πώς γεννήθηκε το μεταναστευτικό. Η Αμερική φέρει ακέραια την ευθύνη για αυτά τα προβλήματα. Άρα και η Αμερική θα πρέπει να κάνει κάτι όσον αφορά τις αραβικές ε, χώρες. Πρόεδρος. Ο κύριος Κασπαρή, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε. 50 εκατομμύρια πιο πολλέ θέσει εργασία από το 2013 έχουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλέ εξ αυτών ε, προήλθαν χάρη στην παγκοσμιοποίηση. Αλλά έχουμε και εκατοντάδε χιλιάδε ανησυχίε στη Χαλιβουργία για παράδειγμα. Και πάλι λόγω της ε, παγκοσμιοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σα παρακαλέσω να χρησιμοποιήσετε και να αξιοποιήσετε το G7 για να μειώσετε του κινδύνου και να αυξήσετε τι ευκαιρίε, για να μπορέσουμε να επωφεληθούμε την παγκοσμιοποίηση και στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α πάρουμε το παράδειγμα τη Κίνα. Έχουμε ένα δισεκατομμύρια εμπορικό όγκο την ημέρα ε, μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα σήμερα. Τεράστιο δυναμικό, τεράστιος προμηθευτής ε, τεράστια αγορά από πλευρά μα. Αλλά λόγω τη Κίνα ακριβώ έχουν δημιουργηθεί θέσει εργασία πάρα πολλέ, αλλά αυτό προκαλεί παράλληλα και ανησυχίε σε πολλού. Α μην τα ισοπεδώσουμε όλα, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά εμπορικές, τομεί, σε ό,τι αφορά τα υποδήματα, για παράδειγμα τη χαλιβουργία τώρα. Σας παρακαλώ λοιπόν αξιοποιήσετε την ευκαιρία του G7 προκειμένου να μιλήσετε με τους διεθνείς εταίρους και να διαμορφώσετε την ε, παγκοσμιοποίηση προκειμένου να έχουμε πιο πολλές θέσεις εργασίας και λιγότερες ανησυχίες. Και τελευταίο, θα ήθελα να έχουμε ανοιχτές αγορές, αλλά θα ήθελα και στο μέλλον να έχουμε και στην επιμηχανία θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν να εργαστείτε προκειμένου οι βιομηχανίε στην Ευρώπη να μπορέσουν να επιβιώσουν και να δημιουργούνται νέε θέσει εργασία στι βιομηχανίε. Ιδάλλον θα καταρρεύσει το μέσα αυτό. Σε ευχαριστώ ο κύριο Ταν για 1,5 λεπτό. Και αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις αρχέ του έτου ε, ο πρόεδρο ε, μετέβησε στην Ευρώπη για να προετοιμάσει το G7 και έχει ένα σαφές μήνυμα λοιπόν προς την Ευρώπη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Σήμερα η Κίνα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και άλλες αναδυόμενες αγορές έχουν ήδη τέτοια προβλήματα. Το G7 αποτελεί παραδοσιακά τη μοναδική μορφή οικονομικού συντονισμού παγκοσμίω. Και το γεγονός ότι απευθύνεται λοιπόν αυτή η έκκληση έχει να κάνει με τον φαύλο κύκλο που έχει ξεκινήσει στην Ιαπωνία. Έχει να κάνει με τις ε, ευρωπαϊκές δυνάμεις, ε, με τον κύριο Σόιμπλε, με τη Γερμανία. Την προηγούμενη εβδομάδα, Η μοναδική απάντηση που έχει να δώσει ήταν ε, μεταρρυθμίσει, τα μεταρρυθμίσεις. Ο Ιάπωνας πρόεδρος όμω έχει δίκιο. Δεν αρκούν οι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει. Οι ευρωπαϊκές αρχέ θα κάνουν πιο πολλά για να τονώσουν τη ζήτηση και πολύ φοβάμαι ότι το G7 θα λήξει με μια θλιβερή, ένα θλιβερό διχασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια προβολή των προβλημάτων που δεν μπορούμε να απειλήσουμε προς τα έξω. Ο κ. Μαριάς, ένα λεπτό. Η διάσκεψη των G7 είναι ανίκανη να δώσει λύσεις στα προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς εμένει στη λιτότητα και συνεχίζει να υποστηρίζει την οικονομία καζίνο σε ένα πολυπολικό κόσμο το αυτάρεσκο σχήμα των g7 δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στη σύγχρονη οικονομία χωρίς να λάβει υπόψη του την ανερχόμενη δύναμη των brics. απαιτείται λοιπόν μια νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική που θα δίνει λύσεις στο πρόβλημα της φτώχειας θα διασφαλίζει μια δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου και θα προωθεί τη διαγραφή του επονίδης του χρέους που καταδυναστεύει τα κράτη. γι' αυτό και δεν εμπιστευόμαστε τα συμπεράσματα που θα βγάλει η επικείμενη διάσκεψη των g7 όσον αφορά το ελληνικό χρέο. Καθώ η χθεσινή απόφαση του eurogroup επιβεβαιώνει ότι οι δανειστέ τη Ελλάδα γδέρνουν το βόδι δύο φορές. αντί λοιπόν η ευρωπαϊκή ένωση και το του να κουρέψουν το ελληνικό δίθεν χρέο και να ρυθμίσουν την εξόφληση του υπόλοιπου με ρήτρα ανάπτυξη όπως έπραξαν ήδη στην περίπτωση τη ουκρανίας τελικά αρνούνται την απομείωση του ονομαστικού χρέου, απαιτούν μέτρα λιτότητα και αδιάκοπη δημοσιονομική προσαρμογή καθώς και διαρκές επί 99 χρόνια ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Κούσο Περμούιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Περίπλοκα τα πράγματα σήμερα. Ε, το, G7, το G7 πώς ε, δημιουργήθηκε. Είναι ε, μια παλιά συσχέτιση δυνάμεων που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 σε ένα πολυπολικό κόσμο και δεν αντιλαμβάνεται ότι είμαστε στο τέλος της δεύτερης παγκοσμιοποίησης. Αυτοί που μας έλεγαν ότι όλη η κυριαρχία του κόσμου πρέπει να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρισκόμαστε λοιπόν στην καμπή ενός πολυπολικού κόσμου και μας το καταδεικνύουν τα γεγονότα κάθε μέρα αναφέρεστε σε παγκόσμια οικονομία και στις ε, προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης ε, και ε, πλήττει την οικονομική ατζέντα που προωθήσατε εσείς και δεν λέει τίποτα για τη δημοκρατική συζήτηση. Αναφέρεστε στο δίκαιο εμπόριο. Επιτρέψτε μου να κανχάσω, διότι πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να βοηθήσουμε τις αναδυόμενες χώρες και τις, τα αίτια της μετανάστευσης. Έχουμε κρίση μετανάστευσης, προσφυγική κρίση και κόσμο νεοφιλελεύθερης ε, κοπής. Για ένα λεπτό ο κύριος Κλένκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον κύριο Τίμερμανς και να τον ευχαριστήσω που μας ε, παρουσίασε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από την 42η Σύνοδο του G7, η οποία ε, καταλήγει σε κοινέ θέσεις για τα παγκόσμια θέματα στα τελευταία χρόνια. Πιστεύουμε ότι οι οικονομικοί δείκτες αυτή τη στιγμή πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση μεν, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε αυτούς ε, στους οποίους δεν έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και ε, Γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διαρθρωτικών Επενδύσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έπρεπε να χρησιμεύσει ως ένα από τα εργαλεία που θα βοηθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των κρατών μελών. Πιστεύω ότι όσον αφορά το G7, πέραν των θεμάτων που αναφέρθηκαν από τον κύριο Τίμερμαντς, ε, πιο συγκεκριμένα λύσεις για τη μεταναστευτική κρίση και άλλα ζητήματα, θα πρέπει να δούμε και ποια θα μπορούσε να είναι η συνεισφορά μου ε, στην επίλυση της μεταναστευτικής κρίσης ε, και πώς μπορούμε να το συνδυάσουμε με τους αναπτυξιακούς στόχους. Επίσης πρέπει να ενισχύσουμε τις εμπορικές σχέσεις, να συνάψουμε συμφωνίες οι οποίες ε, θα λαμβάνουν υπόψη τους τα συμφέροντα των καταναλωτών μας, θα λαμβάνουν υπόψη και τις προδιαγραφές μας και τα πρότυπά μας όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και περαιτέρω συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική επίσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκίλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ε, έχουν αναφερθεί επανειλημμένως εδώ. Τρομοκρατία, μεταναστευτική κρίση, ενέργεια, χρηματική αλλαγή. Και ακόμα προσπαθούμε να ε, ανταποκριθούμε στις συνέπειες της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επομένως, το G7 πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Ζούμε σε έναν διασυνδεδεσμένο, αλληλένδετο κόσμο και πρέπει να βρούμε κοινέ λύσεις. Το G7 αποτελείται από τις πιο ισχυρές οικονομίες του κόσμου και πρέπει να αντιμετωπίσουν τα επίπεδα της ανεργίας που αντιμετωπίζουμε, να αντιμετωπίσουν το θέμα της αύξησης των θέσεων εργασίας. Γιατί μόνο από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις η σύνοδος αυτή ε, σωστά ε, θα ασχοληθεί και με τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου για την παραμονή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί think tank ε, ε, προειδοποίησαν σήμερα ότι εάν επεκταθούν τα μέτρα λιτότητας σε άλλα δύο χρόνια θα μπορέσουμε να έχουμε μας στον προπολογισμό. Αν θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν να πληγούμε όλοι σε παγκόσμιο επίπεδο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αναλάβει τα ενία και να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, διακόπτη πρόεδρο την κυρία Γκίλ, μας ενδιαφέρει κυρίως ε, να μείνουμε και όχι να φύγουμε. Η κυρία Σπινέλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στην ε, ανοικοδόμηση του G8 και την το πολιτικό οικονομικό άνοιγμα προς τη Ρωσία. Θεωρώ ότι πρέπει κατεπηγόντως να ξαναδούμε τις σχέσεις με τις ΗΠΑ εν ώψη του δημοψηφίσματος και των ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και των εκλογών στις Ηνωμένε Πολιτείες. Καλύτερα να τα συζητήσουμε νωρίτερα, να δούμε τι συνέπειε θα έχουμε και με Brexit και με χωρίς Brexit. Όσον αφορά τη Μόσχα, δεν ξέρω αν η Ευρώπη ενδιαφέρεται σε τετραπλάσια στρατιωτική παλουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και των ΝΑΤΟ που θα ε, αποξενώσει ακόμα περισσότερο τη Ρωσία. Η ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα είναι κερδισμένε με τον, ε, με τον Τραμπ ή χαμένε με τη Χίλαρη Κρίντον. Να προετοιμαστούμε σημαίνει ότι θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε αυτέ τι πολιτικέ και να έχουμε και εμεί μια δική μα πολιτική. Από αυτέ τι πολιτικέ ε, δημιουργήθηκαν το Ισλαμικό κράτο, οι πόλεμοι, το προσφυγικό όπω το αποκαλούμε, όταν είναι δικό μα πρόβλημα και δική μα αιτία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοφεράτη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επιμείνω σε τρία στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην ευρύτατη μερίσια διάταξη του G7 και ε, δυστυχώς απουσιάζει και ένα σημείο ε, κατά την άποψή μου αδίκως την ε, φοροδιαφυγή. Η πρόταση του ΩΣΑ είναι μια μικρή πρόταση που δεν επαρκεί. Εγώ πιστεύω και ότι όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις σε πολυμερές επίπεδο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πάμε έτη περαιτέρω. Να έχουμε κάποια πράγματα τα οποία θα είναι δεσμευτικού χαρακτήρα, θα προσδίδουν διαφάνεια και θα επιτρέπουν να έχουμε μια εξέταση αναχώρα σε διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις υπάρχει έλλειψη διαφάνειας. Εμείς δεν μπορούμε να καθόμαστε αδύναμοι ε, να βλέπουμε διαπραγματεύσεις ε, των οποίων δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο, ιδίως όταν αφορούν κοινωνικά, ε, περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα καταναλωτών. Όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις πολυεθνικές, θα πρέπει να τηρήσουμε τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλές φορές η αλυσίδα παραγωγής διαγράφει δικαιώματα που αφορούν τους ανθρώπους, ορισμένες φορές και τα παιδιά. Πιστεύω ότι όλα αυτά δεν είναι πλέον αυτά τα οποία επιθυμούμε. Ευχαριστώ. κυρία, ο κύριος Άσης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας μιλήσω για το ε, ε, διεθνές ε, πολιτικό περιβάλλον. Πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να αποφύγουμε ότι ο ιός του εθνικισμού που βλέπουμε σε μεγάλη κλίμακα στον πολιτικό κόσμο δεν θα μας οδηγήσει σε έναν ιό στις ε, διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι ισχυρές ε, παγκόσμιες δυνάμεις όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνουν μια προσπάθεια για να δημιουργήσουμε ένα πιο ευνοϊκό και διάφανο περιβάλλον για τις εμπορικές σχέσεις από ε, την άποψη όμως και της φορολογίας προκειμένου να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Αν δεν δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις θα επανέλθει ο προστατευτισμός με όλες τους τις ολέθριες συνέπειες. Όσον αφορά τώρα την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το θέμα των προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποπειράθηκε να δώσει μια απάντηση, άλλες φορές καλός, άλλες φορές κακός, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο και να ευαισθητοποιήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο για το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι ε, είναι ευνοϊκέ οι συνθήκε και μπορούμε να θέσουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη του G7. Τώρα παίρνουμε στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑΗ. Δύο συνάδελφοι εγγεγραμμένοι. Γραπίνη. Γραπίνη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κυρία Γραπίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί, λέτε, για το μέλλον. Μάλιστα. Επίσης, είπατε ε, για τις επιδοτήσεις που δεν ε, έπιασαν τόπο. Αναφερθήκατε σε πολλά διαφορετικά ε, ζητήματα και μιλήσατε και για κάποια δισεκατομμύρια και που ξε... τα 45 συγκεκριμένα, που ξέρουμε ότι τα επόμενα θα πιάσουν τόπο. Υπάρχει φοροδιαφυγή, μην ξεχνάτε την υπόθεση των εγγράφων του Παναμά. Ε, είπατε ότι το εμπόριο πρέπει να είναι ελεύθερο. Σωστό είναι αυτό, αλλά πρέπει να είναι και δίκαιο. Έχουμε όλες τις πληροφορίες για να είναι δίκαιο το εμπόριο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα πρέπει να ε, είναι σωστές ε, οι συνθήκες ε, ίσως ο ανταγωνισμός και έχουμε πλήρη πληροφόρηση σε διεθνές επίπεδα. Νομίζω ότι η οικονομία χρειάζεται κανόνες, να είναι ελεύθερη αλλά όχι ασίδωτη. Το εμπόριο να είναι δίκαιο και ελεύθερο. Ευχαριστώ κύριο Σκουτσούκ. Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Τίμερμανς, η σύνοδος G7 στην Ιαπωνία έρχεται στην ε, εύθετη στιγμή, σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων σε όλο τον κόσμο, κρίση νομισματική, τρομοκρατικές απειλές, κλιματικές αλλαγές, πολλές, πολλές περιφερειακές συγκρούσεις, όλα αυτά τα προβλήματα στα οποία πρέπει να δοθούν λύσεις και πρέπει να προσδορίσουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες και δεσμεύσεις. Η σύνοδος του G7 έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να δώσουμε έμφαση στην μεταναστευτική κρίση και την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας, το ελεύθερο εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει έμφαση στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής φοροαπάτης. Πρέπει να αναλάβει και να εκτελέσει τις δεσμεύσεις της ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ τώρα τον λόγο κύριος Τίμερμαντς, παρακαλώ. Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ προς τον ε, αγαπητό κύριο Γκίκολτ που μου επιθύνε δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Θα πρέπει για το πρώτο να σας απαντήσω γραπτός κύριε Γκίκολτ, δεν ε, έχω πρόκειρα τα στοιχεία, για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και τις συγκρούσεις συμφερόντων αυτών. Έγινε επιμακρών συζήτηση και με το Κοινοβούλιο τον κύριο Ντεγιόγκ και άλλους συναδέλφους σας ε, θα κατατεθεί πριν το τέλος του μήνα η σχετική έκθεση της Επιτροπής και θέλω να πω ότι όντως αντιμετωπίζουμε μεγάλες μίσονες παγκόσμιες προκλήσεις τα θέματα που συζητήθηκαν αλλά το να χτίσουμε τώρα αν υψώσουμε τύχη δεν θα μας βγάλει από τα ε, προβλήματα. Μπορεί να είναι σωστό να λέμε να εγκαταληφθούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα το ε, οποίο συζητείτε. Το ελεύθερο εμπόριο θα είναι μια λύση για τις παγκόσμιες προκλήσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημογραφική κατάσταση επίσης. Εάν εμείνουμε σε αυτά που γνωρίζουμε, το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να υπεραμεινθούμε των κεκτημένων μας και το μόνο που θα καταφέρουμε θα ήταν απλώς να επιβραδύνουμε την ύφεση, την υποβάθμιση. Εάν θέλουμε όμως να δώσουμε πραγματικές λύσεις πρέπει να προχωρήσουμε προς μια αηφόρο οικονομία, να ε, ενστερνιστούμε την ψηφιακή οικονομία, να προχωρήσουμε προς μια πιο αποτελεσματική ένωση, κυκλική οικονομία. Αλλαγές δηλαδή. Αλλαγές χρειάζονται με τα απαραίτητα βήματα προς σωστή κατεύθυνση και έτσι μόνο μπορούμε να οικοδομήσουμε επαρκή οικονομική ανάπτυξη που δεν θα ε, καταστρέφει τη γη, θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους και θα οικοδομήσει εκείνο το περιβάλλον που θέλουν κατά τη μέγιστη πλειοψηφία τους οι Ευρωπαίοι για να αντιμετωπίσουμε και τις δημογραφικές ε, προκλήσεις. Αυτό θα προτείνει ως λύση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη G7 το παγκόσμιο εμπόριο να το αξιοποιήσουμε ως ένα μέσον χωρίς να, είμαστε, να έχουμε αφελή στάση απέναντι χρήση των ε, πόρων με μια ευφύ ε, εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων με ευφύης λύσεις. Χρειάζεται να δώσουμε περισσότερη προσοχή και συμφωνώ με όσους το είπαν στην υλοποίηση των συμφωνιών των Παρισίων και αν μπορείτε να παρακολουθήσετε το συλλογισμό μου για μια αηφόρο οικονομία αυτό συνεπάγεται πως πρέπει να επιβραδυνθεί η ε, αύξηση της ε, θερμοκρασίας της γης. Είναι κάτι το οποίο συμφωνήθηκε στο Παρίσι και πρέπει και στο πλαίσιο της G7 στην Ιαπωνία να συζητηθεί. Και κλείνοντα, θα ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά, γιατί ποτέ δεν αρκεί. Η κρίση τη μετανάστευση, η κρίση προσφυγική δεν πρόκειται να πάψουν από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν πρόκειται να εξαλειφθούν με το να τεθεί επιτέλου ένα τέρμα στον πόλεμο στη Συρία. Θα είναι τεράστιες οι δημογραφικές κινήσεις από την Αφρική και άλλες περιοχές του κόσμου και είναι προς δικό μας κεντρικό συμφέρον να εξασφαλίσουμε αηφόρο ανάπτυξη στην ε, γειτονία μας και σε αυτό εννοώ, περιλαμβάνω ολόκληρη την ευρύτερη γειτονία και ολόκληρη την Αφρική. Πρέπει να συστήσουμε θέματα και για τη μετανάστευση και για τις ευκαιρίες και για μια αξιοπρεπή διακυβέρνηση με βάση, με μια σωστή διακυβέρνηση με βάση το κράτος δικαίου, όλα αυτά τα οποία θα γίνουν παράγοντες σε παγκόσμιο επίπεδο για αποφασιστικές επιλογές που θα πρέπει να πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να διαφυλάξουμε και την ευημερία μας ε, ή αδιαφορετικά θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα εισαγάγουμε αστάθεια και φτώχεια από άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτή πρέπει να είναι συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Σύνοδο των 7 ε, ισχυρότερων κρατών. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο, ο Υπουργό κ. Κούντερ εκ μέρου του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς Επιτρέψτε μου να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστερημένη άφηξη κατά τη διάρκεια αυτή τη σημαντική συζήτηση. Ήδη ζήτησα συγγνώμη από τον κύριο Τέλιτσα, τον κύριο Λεμπρετό και άλλου συναδέλφου που δεν του άκουσα. Είχαμε πραγματικά μεγάλη σύγκρουση ε, συμφερόντων λόγω τη επίσκεψη αυτή τη αυτού μεγαλειότητα του βασιλέου. Ε, και θα ήθελα τώρα να απαντήσω στα σχόλιά σας. Όπως είπε ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ηγέτες ε, του G7 θα συζητήσουν διάφορα θέματα παγκόσμια σημασίας, ε, όπου μπορεί πραγματικά να επιδείξει ηγετική στάση η ομάδα των 7. Οι εσωτερικέ και εξωτερικές προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζουμε, είναι αλληλένδετες. Και καλό και σημαντικό είναι να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική συνάντηση η Ευρώπη είναι ε, συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχει εκεί για την αλληλένδετα τα θέματα ασφαλείας, τρομοκρατίας, μετανάστευσης και χρειάζεται συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων μαζί με τους άλλους συναδέλφους ε, της ομάδας των 7. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με ένα θέμα που είναι πολύ ψηλό, όπως γνωρίζετε, στις ε, δικές μας προτεραιότητες. Η κρίση προσφυγική και μεταναστευτική είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα και προκλήσεις και δεν είναι πραγματική δοκιμασία, αλλά και δοκιμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Και έχει πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συζητηθεί στην Ιαπωνία, στην ομάδα των 7, διότι ε, πληττόμεθα πάρα πολύ σοβαρά και οι υπόλοιποι φίλοι ως κατά τα άλλα είναι παγκόσμιο το θέμα και χρειάζεται παγκόσμια απόκριση και αντιμετώπιση. Γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί και ιδέουσα παγκόσμια προσοχή. Ελπίζω να είναι όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα τα πράγματα στο G7. Βέβαια, δεν είναι ο οργανισμός εφαρμοστικός ε, η ομάδα των 7, αλλά μπορεί να καθοδηγήσει, ε, να καταδείξει ότι είναι παγκόσμια η ευθύνη και η ανάληψή της. Και οι ηγέτες μας προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν. η οικονομική μας ενίσχυση και πάλι θα είναι πιο αποτελεσματική αν εγγραφεί σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την προώθηση της ειρήνης, ε, της ασφάλειας και αντιμετώπιση μετανάστευσης. Κοιτάξτε τα θέματα που μας απασχολούν η Συρία αλλά και οι ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή. Άρα αυτό το θέμα ε, με τις μετανάστευσεις δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο. Χρειάζεται διεθνείς ε, λύσεις παγκόσμιες, βεβαίως στα πλαίσια των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Χρειάζεται λοιπόν παγκόσμια απάντηση. Στο G7 θα γίνει αυτό. Είναι ένα προνομιούχο φόρουμ ε, όχι μόνο για αυτά τα θέματα, αλλά για να συσφίξουμε τις σχέσεις μας, για να ε, έχουμε πιο ε, δίκαιο καταμερισμό των ευθυνών και του βάρους. Η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει με πολύ αργούς ρυθμούς, δεν ε, δημιουργούνται αρκετές θέσεις εργασίας και υπάρχει κίνδυνος ε, πραγματικά ύφεσης. Και έχει έρθει η ώρα για τους ηγέτες ε, της ομάδας των 7 να ε, δείξουν ε, ότι δεν είναι μόνο απόλυτη προτεραιότητα μας να επανέλθει η οικονομία, αλλά θα πρέπει ο καθένας να τακτοποιήσει τα του οίκου του, με ευθύνη ο καθένας για τη χώρα του και με συλλογική ευθύνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο G7 έχουν μάθει πολύ ε, το μάθημά του το διδαγμά ότι η απομόνωση, η δημοσιονομική, η φορολογική κτλ. δεν βοηθάει για να ε, αναπτυχθεί η παγκόσμια οικονομία. Είδαμε και τις πρόσφατες ε, κινήσεις και διακοιμάσεις στις αγορές συναλλάγματος. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις και ο ανταγωνισμός δι' αυτού του ε, δρόμου. Ε, έρχομαι τώρα στο τρίτο θέμα από το διεθνέ εμπόριο. Το 2015 οι ηγέτε ε, τη ομάδα των 7 τόνισαν πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο και οι επενδύσει για την ανάπτυξη τη θέση εργασία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Αύριο θα χρειαστεί να ενισχυθεί η πολυμερή εμπορική διάστασης 13 Μαΐου το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την ευρία υποστήριξη ε, στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διάστημα μετά τον Αερόμπι. Η δημόσια εμπιστοσύνη και υποστήριξη για το θέματα του ελευθέρου εμπορίου έχει μειωθεί γιατί ήταν απογοητευτικό το διεθνές εμπόριο τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να ξανακερδίσουμε του ανθρώπου στο πλευρό μας και να εξηγήσουν οι ηγέτε ε, ποια είναι τα ε, πλεονεκτήματα και τα ωφέλη από τις ανοιχτέ οικονομίες χωρίς προστατευτισμό και ε, με πολυμερές και διμερές εμπόριο και αντίστοιχε συμφωνίες επενδυτικέ για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι και να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ίσους κανόνες παιχνιδιού, την πρόσβαση ε, στις αγορές και τις οικονομίες. Βεβαίως θα πρέπει και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες ε, των πολιτών Η κοινωνική προστασία δεν είναι εμπόδιο για το ελεύθερο εμπόριο, το αντίθετο. Θέλω να αναφέρω ακόμα δύο θέματα. Τη φορολόγηση, ε, ε, άλλη προτεραιότητα που έχουμε κοινή με το G7. Τα έγγραφα του Παναμά έδειξαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε παγκόσμια φορολογικά πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πρωτοπόρος ανέκαθεν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής και της επιθετικής φορολογικής ε, πολιτικής και φορολογικού σχεδιασμού. Έχουμε την οδηγία για την καταπολέμηση του ξεκλήματος του χρήματος για να ξέρουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι και σήμερα το Συμβούλιο ενέκρινε μετά από ε, τη δική σας πρόταση την οδηγία ε, για ε, τη διοικητική συνεργασία σε ό,τι αφορά την εκθέσεις αναχώρα για τα κέρδη των επιχειρήσεων. Επίσης, έχουμε και μια εξωτερική στρατηγική που καλούμε να συσταθεί μια μαύρη λίστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη που δεν συνεργάζονται και το ΕΚΟΦΗΝ εργάζεται προς μια κατεύθυνση γενικής αντιμετώπισης της οδηγίας για την ε, φοροδιαφυγή, και τη φοροαποφυγή. Ε, ελπίζω να υπάρξει κάποια φιλοδοξία και μεγάλη σε αυτό το τομέα επίσης. Κατά πολέμηση δημοκρατίας τώρα. Ε, είναι αναπόφευκτο. Ε, ε, ε, αυτό το θέμα κάθε μέρα κάθε φορά μάλλον που υπάρχει μια δεχτή τέτοια τρομοκρατική επίθεση, ένα απεχθέ έγκλημα επηρεάζει όχι μόνο όλη μας αλλά και την ίδια τη ζωή μας και την ποιότητα. Από την περασμένη φορά, την περσινή, συνεδρίαση έχει μειωθεί η επικράτεια που ελέγχει το ΙΣΙΣ και στο Ιράκ και στη Συρία γιατί υπάρχει μαζική πίεση διεθνής από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τους εταίρους μας Βλέπουμε όμως να αυξάνονται οι επιθέσεις ταυτόχρονα, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Ε, η σύνοδος κορυφής των 7, λοιπόν, δεν θα καταγράψει απλώς τα μέτρα, αλλά θα εξετάσει ε, τι ε, επιπλέον θα μπορούσε να γίνει και ελπίζουμε ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της δημοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού να εγκριθεί και να ενισχυθεί η διεθνή συνεργασία κατά αυτών των απειλών και να γίνει όσο γίνεται περισσότερο αποτελεσματική. Στη συνέχεια θα συζητήσουν οι ηγέτε γενικότερα την κατάσταση στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη, αλλά και την Ουκρανία. Θα πρέπει οπωσδήποτε ε, οι συμφωνίε του Μίνσκ να ε, υλοποιούνται στο ε, ακέραιο και όλα τα μέρη να την στερνιστούν αυτή την προσπάθεια. Αυτά. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το θέμα του G7 θα πρέπει να διευρύνουμε την διεθνή κοινότητα των ε, εθνών και των κρατών που μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες και είναι προσιλωμένα στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πάρα πολύ σημαντική είναι και η αλληλεγγύη και ε, η πρόθεση μιας διεθνούς τάξεως που να βασίζεται σε κανόνες. Αυτά είναι άλλωστε και η συνθετική μας ε, κρίκη στην Ευρώπη και κάτι που διέπει το δικό σας έργο εδώ και τις εργασίες του Κοινοβούλου προσβλέπω ε, στη συνάντηση αυτή των 7 και σας ευχαριστώ και πάλι για τη σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ.